Ωραία συνάδελφοι, θα περάσουμε απευθείας στις ψηφοφορίες. Αλλά πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, έχω κάποιες ανακοινώσεις για τους συναδέλφους της ΔΕΒΕ, τις οποίες θα διαβάσω. Η πρώτη είναι ψηφοφορία για τις συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες με το Βιετνάμ αναβάλλεται. Γιατί η ΙΝΤΑ επίσης ανέβαλε την εργασία της για το θέμα αυτό επαόριστον, γιατί υπάρχουν θέματα στο Συμβούλιο. Δεν θέλαμε να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση ΝΤΕΒΕ εάν ε, δεν γνωρίζουμε πότε θα έχουμε την επίσημη υποβολή στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές. Ίσως να είναι μετά τις εκλογές. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι την επόμενη Τρίτη 12 Φεβρουαρίου έχουμε Διεθνή ημέρα κατά, κατά των ε, παιδιών ως στρατιώτες. Είναι η λεγόμενη ημέρα των ε, ματωβαμένων χεριών. Είναι η μέρα κατά την οποία θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν ε, κρίσεις όπως το Μιανμάρ, τη Συρία, τη δημοκρατική, την, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στρατιώτες. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το αποτρόπαιο φαινόμενο που ε, καταστρέφει τη ζωή των παιδιών που δεν πρέπει να συμμετέχουν σε σειράξει. Τρίτον, έγκριση των αποφάσεων και στάσεων των συντονιστών. Οι αποφάσει για τις 22 Ιανουαρίου είναι στα εγγραφά σα Αν δεν υπάρξουν σχόλια μέχρι το τέλο της συνεδρία, θα θεωρείτε ότι είναι Τέσσερα. Η Επιτροπή δεν θα κάνει καμία ανακοίνωση. Άρα δεν θα μα κάνει καμία ανακοίνωση. Η Επιτροπή έχει αποχωρήσει. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Το 7 πέρασε, ε, αναβάλλεται, το 8 αναβάλλεται, το 9 αναβάλλεται, το 10 αναβάλλεται. Η πρώτη ψηφοφορία είναι το 11. Ναι, τον Αντέλα. Ωραία. Ψηφίζουμε τώρα για το 11. Η χρηματοδότηση, επιτήρηση και διαχείριση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Σας παρακαλώ. Υπάρχει πολύς χώρος έξω άμα θέλετε να μιλήσετε. Μαρία, σημαντικό θέμα. Γι' αυτό να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους κοιόδης. Και αυτό ισχύει για τις τρεις ψηφοφορίες που θα κάνουμε τώρα, 11, 12 και 13. Κάναμε κάθε προσπάθεια από κοινού για να επιτύχουμε συμβιβασμούς και για να δώσουμε μια καλή γνωμοδότηση για τη γεωργική πολιτική ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η γεωργία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμη ανάπτυξης. Χθες το βράδυ ε, συζητήσαμε ακόμη για ε, συμβιβαστική λύση. Για το σημείο 12 θα υπάρξει προφορική τροπολογία από πλευρά του ΕΛΚΑ, την οποία στηρίζω. Χαίρομαι που μέχρι τελευταία στιγμή αγωνιστήκαμε για να βρούμε μια κοινή λύση. Ευχαριστώ οσου συμμετείχαν και τους συνεργάτες μας που επίσης εργάστηκαν σκληρά για τα θέματα αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έλλη, θες να ρωτήσει κάτι. Ε, ναι, βρίσκω την κάρτα μου. Μπορώ να ψηφίζω ε, δια ανατάσσεως της χειρός. Ναι, αλλά αν είναι αποφασιστική η ψήφος δεν θα μετρήσει. Αυτός ο κανόνας. δηλαδή η ψήφος σας θα αλλάζει το αποτέλεσμα είναι συνεργάτη σα δεν μπορεί να πάει να την πάρει το γραφείο σα. Μα πάντα έχουν και μία ε, δεύτερη κάρτα. Α πάει κάποιο από το γραφείο σα να την βρει. Η Αν Μακλόχλιν, η προηγούμενη βηματάρχη μας, ε, θα είναι αρμόδια τώρα για τις κάρτες. Στείλτε κάποιον να πάρει μια τέτοια δεύτερη κάρτα. Ωραία. Δεν κάθεστε ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες, οπότε θα υπάρξουν δυσχέρειε. Νόιζερ επικεφαλή των ε, σοσιαλιστών και ο κύριος Γίγκολ για, τους, ε, για το ΕΛΚ. Εντάξει, ωραία. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουν 62. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ. Ω, λάθος, λάθος, καταπίπτει. 19 υπέρ, κατά αποχές. Δεκτή. 71 υπέρ, κατά αποχές. Δεκτή. 20, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 8-13. 72 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 73. Δύο τμήματα. Τρία τμήματα. Όχι, δύο τμήματα. Α, με μπέρδεψαν τα τρία συν στο κατάλογο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Ναι, περίπου ίδιο σχετισμός. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 21. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 75. Υπέρ. Κατά. Α, να ελέγξουμε την 21. Καλώ. Ελέγχουμε τον 21. Άρχεται. Συγγνώμη, νόμιζα πω το ΕΛΚ ήταν υπέρ. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πέρα. Ισοψηφία 10. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχέ, Δεκτή. 76 υπέρ. Κατά απόχέ, Δεκτή. Συμβαστική ήττα υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πιστεύω αλλά την ελέγχουμε την 81 έρχεται, πέρας Α, περνάει με 11-10. 24 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, μισό, δεν βλέπω. Παρακαλώ, υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ. <clears throat> κατά αποχές ελέγχουμε. Την 82. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11-10. Αιτιολογικέ σκέψεις. Ε, συμβαστική α, υπέρ. Ναι. Εάν αλλάζει το αποτέλεσμα, τότε δεν μετράει. Πρέπει να γίνει με κάρτα. Αυτός είναι ο κανόνα. Άρα, Έλλη, χρειάζεται η κάρτα σου. Αν θέλετε να μπορέσετε να ψηφίσετε για τις ε, σημαντικές. Λοιπόν, συμβαστική α, η αιτιολογική σκέψη έχουμε περάσει. Υπέρ κατά αποχές, δεκτή. Α, έχετε κάρτα, ωραία. <clears throat> συμβαστική β, υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχέ. Δεν είδα τι ψηφίζουν οι σοσιαλιστές. Δεν είπατε. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε την 36 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή Μα το έλκυνταν υπέρ 44 δεν ήτανε Α Καλά. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια σύγχυση, γι' αυτό ας ελέγξουμε Τις 44 άρχεται. Συγγνώμη. Πέρας. Δεκτή, 13-9. 46 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 κατά τμήματα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ελέγχουμε ελέγχουμε το δεύτερο μήνα της 7 είναι πιο εύκολο όταν οι πολιτικές ομάδες κάθονται μαζί πέρας απορρίπτεται Ναι, τι θα γίνει, τι γίνεται όμως αν εγκριθεί τμήμα τις προηγούμενες. Καλά, α την ψηφίσουμε για να δούμε. 51 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Τη 60 άρχεται. Τώρα, τώρα, τώρα Ελέγχουμε την 60. Ψηφίσατε όλοι. Επί 60. Πέρα. Απορρίπτεται. 10-11. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12. Α, όχι, καταπίπτει. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 26 πρέπει να την ελέγξουμε. Άρχεται. Ελέγχουμε την 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Σοψηφία 10 υπέρ 10 κατά. Τελική τροποποιηθήσα, ε, ε ψηφορία επί του κειμένου ονομαστική άρχεται. Μπορείτε να ανοίξετε παρακαλώ κύριε τεχνικέ την, ε, το μηχάνημα για την τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ και 2 αποχές. Συγχαίρουμε τη Μαρία. Περνάμε στην επόμενη έκθεση της Μαρία, σημείο 12. Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της κοινή γεωρικής πολιτικής και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωρικό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Θέλεις κάτι να πεις για την έκθεση? Όχι, μίλησες πριν για όλες. Πολύ ωραία. Έτσι είμαστε αποτελεσματικοί. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται». «133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται». 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 24 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12 προς 10. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε την 31. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η συμβαστική. Η 37 και η 139. Περνάμε στην 143. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 11 με 11. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, νόμιζα πως το τόλικ είναι υπέρ. Θα ελέγξουμε την 147. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλά κάνετε και ρωτήσατε και ζητήσατε έλεγχο. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος την 152 άρχεται πέρας απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε την 161. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 162. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 11 ψήφους υπέρ, 10 κατά. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της 164. Πέρας. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Α, καταπίπτει και αυτή. Εκατόν εξήντα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το δούμε. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται λοιπόν. 169. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά ελέγχουμε την 177. Πέρας. Εγκρίνατε. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 182 πέρας απορρίπτεται 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε την 184. Πέρας. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές έλεγχο στην 55. Πέρας. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 58. Απορρίπτεται για κάποιο λόγο. 193 υπέρ, κατά, αποχές, συγκρίνεται. 194 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφασαν όλοι. απορρίπτονται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Α, έλεγχος για την 59. Νομίζω ότι πέρασε ότι άρχεται ο έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. 196 άρχεται. Πέρας. 12-10 εγκρίνεται. Σημαντική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ...65 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος για την 65 άρχεται. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται 12-10. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά απόχέ, νομίζω ότι απορρίπτεται έλεγχος για την 67 άρχεται πέρας απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε τελικές σκέψεις 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 79 άρχεται πέρας απορρίπτεται με τεράστια διαφορά δύο υπέρ κατά υπέρ μάλλον συγγνώμη γιατί δύο έλκ δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα κατά αποχές έλεγχος για τη δύο στην αρχή να σηκώνετε το χέρι, να σας προλαβαίνω, να σας βλέπω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-10. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 94 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Όχι. 94 πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Η φιλελεύθερη είναι καθοριστικός το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές το ίδιο 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 101 έρχεται πέρας απορρίπτεται κατά τμήματα για την 8. 8 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα έρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος 102 άρχεται. για την 102 πέρας εγκρίνεται με 11-10. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 καταπίπτει. Α, 107. 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 καταπίπτει 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές ποιες έλεγχος για 14 έρχεται νομίζω ότι απορρίπτεται έλεγχος πέρας εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά έλεγχος 116 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος του πρώτου τμήματος. Άρχεται. Ψηφίσατε πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Α, καταπίπτει. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 123 υπέρ, κατά αποχές 123 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πλησιάζουμε, πλησιάζουμε. Στο τέλος. 125 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος την 127 έρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές 129 υπέρ κατά εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ η διερμηνία θα δεκοπεί τώρα λόγω λήξης του ωραρίου εργασίας των διερμηνών.